Okay, friends. Uh, uh, Αγαπητοί φίλοι, να σας ε, πω λιγάκι πώς θα προχωρήσουμε σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη. Θα, θα ξεκινήσουμε με την ανταλλαγή ε, απόψεων για την έκθεση μπάλας για το κοινωνικό dumping στις 11 και 4 στην αίθουσα PHSC50 ε, θα υπάρχει κοινή συνεδρίαση ε, για την οικονομική ανισότητα και στις 3 θα επανέλθουμε σε αυτή την αίθουσα και θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο Κατάιναν. Ελπίζω να υπάρχουν αρκετοί ε, στην αίθουσα γιατί πραγματικά είναι πρόβλημα όταν προσκαλούμε αντιπρόεδρο και άλλους εκπροσώπους και τελικά βρισκόμαστε πολύ λίγοι στην αίθουσα. Μετά τον κύριο Κατάινεν θα υπάρχουν ψηφοφορίες και μετά από τις ψηφοφορίες υπάρχει ένα νέο σημείο στην ημερήσια διάλαξη. Είναι η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής με τον κύριο Σόγκρος εισηγητή και μετά θα υπάρξει η συνέχιση της κανονικής ημερήσιας διάταξης με τις μικρές επιχειρήσεις ε, μεταφορών και τις ε, πολιτικές απασχόλησης. Έχουμε τις εξής γλώσσες ε, Εκτός από τα ε, κροατικά, ε, το... και κελτικά, ε, έχουμε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες. Στη μία ε, δεν θα έχουμε όμως εστονικά, μαλτέζικα και κελτικά. Και στη συνέχεια εκτός από τα κροατικά και τα κέλτικα θα έχουμε πάλι όλες τις γλώσσες. Εγκρίνονται τα σημεία της μερίσιας διάταξης για τις 24 Μαΐου, ναι. Οπότε συνεχίζουμε με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Γκυγιόν Μπάλας. Merci, Madame la, la Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα πρώτα απ' όλα να πω γιατί ζήτησα αυτήν, ε, τις τροπολογίες, τις συμβιβαστικές επειδή η συζήτηση σχετικά με την έκθεση αυτή είναι ίσως πάρα πολύ μακρά, ε, ο αριθμός των τροπολογιών είναι πολύ μεγάλος, ε, πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά το θέμα είναι λεπτό, όπως ξέρουμε, στις συζητήσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Μου φάνηκε λοιπόν σημαντικό να έχουμε ένα ενδιάμεσο σημείο πρωτού οριστικοποιήσουμε αυτή την έκθεση για μια ψηφοφορία τον Ιούλιο στην Επιτροπή και αν είναι θετική η ψηφοφορία στην Ολομέλεια από το Σεπτέμβριο. Το πρώτο σημείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω ε, δεν είναι. σημαντικό, ε, η, ο τύπος είναι σημαντικό στη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και όδης συγητές με τους οποίους συνεργάστηκα για το θέμα αυτό, διότι έδωσαν πάρα πολύ χρόνο, αφιέρωσαν πολύ χρόνο, ε, συνέβαλαν πάρα πολύ στη συζήτηση. Δεν είχαμε μικρές τυπικές συζητήσεις, εξετάσαμε ενδελεχώς το θέμα. Θέλω να τους ευχαριστήσω διότι μένα από τους δε μαθαίνουμε πολλά παρόλο που έχουμε διχογνωμίες αρχικά και δεν είναι εύκολο να τις ε, υπερβούμε αλλά είναι μια μέθοδος όπου ο καθένας ε, προσφέρει με τρόπο ειλικρινή αυτό που έχει να προσφέρει για να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα συμβιβασμό. Πού βρισκόμαστε σήμερα, κατά τη γνώμη μου βεβαίως μετά το, το άθροισμα των τροπολογιών που κατατέθηκαν, ε, μια ε, μακρά εργασία για να έχουμε συμβιβαστικές τροπολογίες, ένα πρόγραμμα καθιερώθηκε. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάθε συμβιβαστική τροπολογία να συγκεντρώσουμε το σύνολο των ομάδων, να τις αντιπροσωπεύσουμε, διότι πρέπει να διαλέξει κανείς ένα σημείο ανάμεσα στο να μην μπει τίποτα και να περιλάβει όλους για να μπορέσουμε να πούμε κάτι. Υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, όμως υπάρχουν θέματα θετικά στη συζήτηση που είχαμε. Το πρώτο είναι η ικανότητα που είχαμε για μια πλειονότητα των ομάδων, όχι το σύνολο, λυπούμε, δεν μπορέσαμε να έχουμε όλες τις ομάδες παρά μόνο μερικές, αλλά σήμερα είναι οι περισσότερες για το θέμα του ορισμού του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ήταν ένα διακύβευμα σημαντικό, διότι ξέρουμε ότι εκεί βρίσκονται τα προβλήματα, εντοπίζονται τα προβλήματα και οι διαφορές που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στις ομάδες και ανάμεσα στις χώρες. Και αυτός ο ορισμός του dumping δεν μπορούσε να σταματήσει ε, σε κάτι το μονοδιάστατο, γι' αυτό τονίσαμε την σημασία και στον κοινωνικό τομέα, αλλά επίσης και τον αντίκτυπο στον οικονομικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Σχέδιο ε, τροπολογιών συμβιβαστικών μας επέτρεψαν να προοδεύσουμε σχετικά με το θέμα του ελέγχου σήμερα της εφαρμογής ε, των νομοθεσιών των υφισταμένων από κοινωνική απόψεως για να ε, αγωνιστούμε καλύτερα κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ. Νομίζω ότι αυτό ισχύει κυρίως με τις υπενθυμίσεις, ε, τις συνενετικές ε, του σεβασμού των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τηρεί όλους αυτούς τους κανόνες και αυτό είναι μια προϋπόθεση, ένα προαπαιτούμενο, αλλά χρειάζεται και η βελτίωση των επιθεωρήσεων των πραγματικών, των οριζοντίων σχέσεων ανάμεσα στις εθνικές επιθεωρήσεις, τους τρόπους για να μπορούν να αποδώσουν καλύτερα σχετικά με τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Σκέφτομαι τη μετάφραση, τις ανταλλαγές στο νομικό τομέα και επίσης προχωρήσαμε. Ήταν μια μακρά συζήτηση, δύσκολη, επίπονη, διότι έπρεπε να πούμε τι έπρεπε να γίνει και όχι να αφήσουμε εσφαλμένες ιδέες ε, να επιβληθούν, αλλά επιμείναμε πάνω στην ιδέα ότι χρειάζεται μια πολυεθνική συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχυμένη με την θέσπιση των task force ε, πολλήπλευρων ομάδων εργασίας που θα περιλαμβάνουν επιθεωρητές εθνικούς για θέματα συγκεκριμένα και κυρίως ε, ε, για να μπορέσουν να εντοπίσουν τις εταιρείε μαϊμούδες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Μεταφορών με την οποία εργαστήκαμε ε, καλά. Στην αρχή δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο για να βρούμε μια συμφωνία για αφενός αυτό που θα μπορούσε να ενταχθεί ή όχι ανάλογα με τις αρμοδιότητες των δύο επιτροπών και μέσα στην Επιτροπή Μεταφορών, όπου υπήρχαν ορισμένες προτάσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ, είναι σημαντικές αυτές οι προτάσεις και θα τις εντάξουμε αυτές καθεαυτές στην ε, δική μας Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αν το αποφασίσετε στην ψηφοφορία. Είχαμε μια ευρεία ε, συμφωνία μεταξύ των ομάδων. Επίσης προοδεύσαμε για ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα. Πρόκειται για το θέμα της ψηφιακής ε, οικονομίας. Η ψηφιοποίηση επανατοποθετεί με τρόπο διαφορετικό την έκθεση για την κοινωνική προστασία, δηλαδή τη σχέση με την επιχείρηση, το θέμα της σχέσεως εργασίας, τι είναι να είναι κανείς εργοδότης και εργαζόμενος και κάναμε νομίζω προτάσεις χρήσιμες προς την κατεύθυνση άλλων εκθέσεων που ψηφίστηκαν προηγουμένως και πάνω στις οποίες μπορέσαμε να βασιστούμε. Παρ' αυτά παραμένουν σήμερα σημεία τα οποία ε, δεν εγκρίνονται από πλειονότητα των ομάδων και χρειάζεται περισσότερη πρόοδος και περισσότερη εργασία. Το μερικά σημεία και μετά θα περάσω στο σφιαστικό, αλλά τα πρώτα σημεία αυτά δεν είναι αμεληταία, είναι το θέμα ε, της διακοπής παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης της νομοθεσίας κυρίως όσον αφορά τους αποσφασμένους εργαζόμενους. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση που είναι ιδιαίτερη και που απαιτεί όλη την προσοχή μας. Εγώ προσωπικά εκπλήσωμαι στην Ευρώπη ενώπιον της συλλογικής μας ανικανότητας, δεν μιλάω για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, διότι συλλογικά είμαστε ανίκανοι να βρούμε κανόνες ελάχιστους εναρμόνισης για ορισμένα θέματα και βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες μονομερείς αποφάσεις σήμερα και όταν λέω σήμερα, ακόμη και πρόσφατα, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει ορισμένες διαδικασίες απέναντι στα κρατημένη, ορισμένες προσφυγές στη Γερμανία και τη Γαλλία. Δεν νομίζω ότι οι μέθοδοι αυτές, δηλαδή τα μονομερείς αποφάσεις που θα αμφισβητηθούν από την Επιτροπή και μετά θα τροφοδοτήσουν ένα, μια συζήτηση πολιτική πολύ ε, κακή, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να προχωρήσουμε για ορισμένα θέματα σχετικά με αυτήν την διακοπή παροχής υπηρεσιών από τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση σοβαρής ε, παραβίασης είναι δυνατή σε χώρες που την εφαρμόζουν και υπάρχουν σήμερα δύο χώρες που δεν την εφαρμόζουν. Η ιδέα ήταν να γενικεύσουμε την δυνατότητα να γενικεύσουμε ακόμη και την γνωμοδότηση ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεθόδους κοινέ για να υποχρεώσουμε τις ε, επιχειρήσεις να προσέχουν, δεν πρόκειται να ε, τους επιβάλλουμε μέτρα γραφειοκρατικά που δεν μπορούν να διαχειριστούν, να, να προσέχουν στις υπεργολαβίες, ποιες είναι οι επιπτώσεις για τους εργαζόμενους και βεβαίως στις ε, θηγατρικές τους που είναι της δικής τους ευθύνης, θα έλεγα. Το σημείο, τα σημεία ε, διαφορών τα σημαντικότερα είναι για δύο παραγράφους που πρότεινα ως συμβιβαστικές τροπολογίες που έχουν εγκριθεί από ορισμένε ομάδες, μεγάλο αριθμό ομάδων, αλλά όχι μια σημαντική πλειοψηφία. Είναι το θέμα το, της, ε, της εργασίας των αποσπασμένων, της απόσπασης. Εκεί υπάρχει ένα σημείο μεθόδου που θα πρέπει να εκτιμήσουμε. Υπάρχει Υπάρχουν οι προτάσεις της Επιτροπής που τέθηκαν επιτάπητος πρόσφατα. Υπάρχουν αντιδράσεις από διάφορα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Το γνωρίζουμε. Υπάρχει μια έκθεση που ανατέθηκε επίσημα σε δύο ε, η κυρία Μρονσαρτιέ Σαρτιέ από το ΕΛΚ και τη από τις, την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας δεν πρόκειται να προκαταλάβουμε την εργασία που θα γίνει τότε και που θα είναι μια επίπονη εργασία. Ωστόσο, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο ε, για ένα μέρος ε, από εμά, ενώ ξέρουμε ότι η αποσπασμένη εργασία είναι ένα θέμα λεπτό, ευαίσθητο και εκεί όπου το κοινό βλέπει ότι υπάρχει το πρόβλημα του dumping social, του κοινωνικού dumping ως το σημαντικότερο, να μην ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Γι' αυτό για την ώρα μου φαίνεται δύσκολο να δεχθούμε το αίτημα, να δεχθώ το αίτημα που μου υποβλήθηκε να μην έχει υπάρχει τίποτα για το θέμα αυτό των αποσπασμένων στην έκθεση πρωτοβουλίας, θα νομίζω ότι μάλλον θα έπρεπε να έχουμε μια συζήτηση για αυτές τις συμβιβαστικές τροπολογίες για να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε μια συμφωνία γενική και θετική μεταξύ μας. Γιατί, διότι νομίζω ότι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να ψηφίσει μια έκθεση πρωτοβουλίας καταπολέμησης του κοινωνικού ντάμπινγκ και η αποσπασμένη εργασία δεν καλύπτεται για να καλυφθεί αργότερα πολιτικά οι συμπολίτες μας ε, θα ε, είναι πάρα πολύ σκεπτικοί και θα σκεφτούν ότι δεν παίζουμε το ρόλο που θα έπρεπε να διαδραματίσουμε. Η έκθεση πρωτοβουλίας υπάρχει για ε, να διαδώσει ορισμένες ιδέες πάνω στις οποίες πρέπει να βασιστούμε. Δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό, αλλά μια βάση εκκίνησης η κυρία Τίσαν της Επιτροπής έδωσε τη γνώμη της και μετά ε, την διαδικασία ε, της Επιτροπής πρέπει να συνεχίσουμε και το Κοινοβούλιο με γενικό τρόπο χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες και να μπορέσει να δώσει κάτι το θετικό. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Αυτές είναι οι πρόοδοι που είναι ουσιαστικές και ενδιαφέρουσες, αλλά ακόμα έχουμε δρόμο να διανύσουμε και θα έπρεπε να τον καλύψουμε, διότι νομίζω ότι σήμερα αυτός είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καλύψει πλήρως αυτό το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ για να απαντήσουμε στα ερωτηματικά των συμπολιτών μας. Δεν ήθελα να υπενθυμίσω το περιεχόμενο το συζητήσουμε, αλλά βλέπουμε σήμερα ότι το θέμα της αθέμη, του αθέμητου συναγωνισμού, ανταγωνισμού μέσα ε, στην εσωτερική αγορά ε, τροφοδοτεί πάρα πολλές ιδέες ε, και φαντασιώσεις. Θα έπρεπε λοιπόν να παίξουμε το ρόλο μας. Ευχαριστώ, κύριε Ευχαριστώ κύριε Μπάλλα. σκληρή. Uh, το θέμα είναι να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα αποτελέσματα. Θα δώσω το λόγο στη σκιώδη συγγήτρια. Η κυρία Γιασλοβιέσκα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Μπαλάς και το σύνολο της ομάδας του έχουν κάνει μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ και ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίσατε και ο τρόπος που ακολουθήσατε για να καταλήξετε στις συγκεκριμένες τροπολογίες ήταν πολύ καλός. Χρειάστηκαν 20 συναντήσεις για να πετύχουμε τη σύγκληση αυτή. Πάντως οι εργασίες μας στα πλαίσια του κοινωνικού ντάμπινγκ πλησιάζουν στο τέλος τους και ε, υπάρχουν κάποια θέματα βέβαια πάνω στα οποία δεν έχουμε ακόμα μία κάποια συμφωνία. Αρκετά είναι τα μέλη που έχουν κάνει κριτική σε, στο θέμα της έλλειψης μιας επίσημης, ενός επισήμου ορισμού του κοινωνικού ντάμπινγκ. Δεν έχουμε δηλαδή ένα όρο ο οποίος να έχει ξεκαθαρή νομική ισχύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήταν χρήσιμο. Οι περισσότερες πολιτικές ομάδες θεωρούν ότι στην ουσία είναι στρεβλές πρακτικές οι οποίες έχουν σαν στόχο να παρακάμψουν τον νόμο και αυτό είναι το dumping και στον τομέα τον κοινωνικό. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα όμως στις πολιτικές ομάδες. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν μπορεί να υποστηρίξει όλες τις συμβιβαστικές, ιδιαίτερα σε θέματα όπως το δεσμευτικό σύστημα καταγραφής των αποσπόμενων εργαζομένων Ε, το θέμα του τερματισμού της παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση ε, παραβίασης της νομοθεσίας για τους αποσπόμενους εργαζομένους, ε, το θέμα του τομέα του, των αερομεταφορών που είναι κάτι που ανήκει στην Επιτροπή Μεταφορών, η σχέση ανάμεσα στα οικονομικά και στα κοινωνικά δικαιώματα, όπως και το LA νέο και το M, συμβιβαστικές LA νέο και M για την μεταρρύθμιση της οδηγίας για τους εργαζομένους αυτούς. Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν πρέπει να μπούμε σε επίπεδο λεπτομέρειας. Θα πρέπει οι αρμόδιοι εισηγητές που έχουν καθοριστεί να προχωρήσουν στις προτάσεις αυτές. Να θυμίσω ότι το κοινωνικό dumping δεν είναι κάτι το οποίο περιορίζεται μόνο στο θέμα της ε, απόσπασης εργαζομένων. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο γενικό σαν πρόβλημα. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σαν παράδειγμα στην παράνομη εργασία, στις εταιρείες γραμματοκιβώτια, στην ε, άσκηση βίας για εργασία, προς εργασία, και στην, στον σεβασμό της αρχής ίσης αμοιβής για ίση απασχόληση. Νομίζω λοιπόν ότι κάποια άλλα μέτρα τα οποία προτείνονται θα μπορούσαν στις διάφορες χώρες μέλη να υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ που προσθέσατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, λέει η κυρία Ντλαμπάγιοβα. Ευχαριστώ τον κύριο Μπάλας και τους Σκιώδης. Είχαμε μαζί του εξαιρετικές, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις. και η κυρία Γιασλοβέσκα και ο κύριος Μπάλας ε, έκαναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να λειτουργήσω λίγο θεωρητικά, λίγο φιλοσοφικά και να κάνω τρεις τα επιπλέον παρατηρήσεις. Καταρχάς θα ήθελα να σχολιάσω το γενικό μήνυμα το οποίο εκπέμπει η συγκεκριμένη έκθεση. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ικανοποιημένη για την γενική τάση και το μήνυμα της έκθεσης επαναλαμβάνει σε πάρα πολλά σημεία και πάρα πολύ συχνά το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων σαν βασική αιτία κοινωνικού ντάμπινγκ. Ενώ δεν αποτελούν παρά μόνο το 1% της, του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. Είναι μια έννοια η οποία συνδέεται με κάθε μορφή παράκαμψης νομικών ρυθμίσεων για να μειωθεί το εργατικό κόστος είναι η ε, δραστηριότητα αυτή ε, της απόσπασης εργαζομένων μια νόμιμη δραστηριότητα και αν υπάρχουν καταχρήσεις θα πρέπει αυτό να γίνει μέσω της εφαρμογής των κανόνων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. Δεν απαιτούνται νέες συνεχώς ρυθμίσεις. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις καταχρήσεις ενισχύοντας επίσης σε διεθνές επίπεδο και τις ε, εργασιακές επιθεωρήσεις, τις επιθεωρήσεις στους τόπους εργασίας. Ο σεβασμός των κανόνων δεν μπορεί να ονομαστεί άδικος και δεν μπορεί να ονομαστεί επίσης κοινωνικό ντάμπινγκ. Το θέμα λοιπόν της ανταγωνιστικότητας ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διατηρηθεί στην Ευρώπη και να μην ανασχεθεί από προστατευτικά μέτρα, γιατί αυτό θα στερήσει από την Ευρώπη ένα καλύτερο μέλλον. Στην έκθεση μερικές φορές κρυφόμαστε πίσω από το θέμα της απόσπασης, κρύβουμε μάλλον κάποια άλλα θέματα της αγοράς εργασίας που αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες πολύ σοβαρά. Δεν θέλουμε να τα συζητήσουμε, δεν θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε και κρυβόμαστε πίσω από το θέμα της απόσπασης. Ε, το να υποστηρίζουμε επίσης θέματα για τα οποία δεν υπάρχουν αποδείξεις αλλά βασίζεται ο εισηγητής μόνο σε συναισθήματα είναι κάτι το άδικο για τους ίδιους τους εργαζομένους. Στην ουσία η απόσπαση των εργαζομένων χρησιμοποιείται σαν αποδιοπομπαίος τράγος για το κοινωνικό ντάμπινγκ. Δυστυχώς δεν υπάρχει παρά ένα μικρό ε, ένα μικρό κομμάτι της έκθεσης το οποίο αναφέρεται σε θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε τώρα. Για την αρχή ίση αμοιβή, ίση απασχόληση είναι μια βασική αρχή στον ίδιο χώρο. Είναι ένα ωραίο σύνθημα το οποίο δεν έχει τίποτα να κάνει με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην Ευρώπη και ψευδόμεθα όταν λέμε ότι τις διαφορές αυτές μπορούμε να τις καταργήσουμε σήμερα. Για να τις καταργήσουμε θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια, όσα χρόνια ξοδέψαμε και εμείς συζητώντα το θέμα αυτό. Οι διαφορές αυτές μπορεί να οφείλονται σε ιστορικές, ε, θα έλεγα, διαφοροποιήσεις, έχουν προκληθεί από την πραγματικότητα που επικρατεί σε κάθε χώρα και δεν θα πρέπει η ιστορία να επαναλάβει τον εαυτό της. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν παραδείγματα πως οι εργαζόμενοι ε, να ε, ανήκουν ε, σε διαφορετικά συστήματα και συμβάσεις ε, τις οποίες υπογράφουν σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που επικρατούν και στην Ευρώπη, που υπάρχουν και στην Ευρώπη και σε χώρες εκτός Ευρώπης. Η διαφορετικότητα αυτή είναι κάτι το θετικό και πρέπει να μας ενώνει. Θα ε, έλθω τώρα στο τέλος στον ορισμό της, του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ο ορισμός που προτείνεται είναι πάρα πολύ μακρύς είναι πάρα πολύ περίπλοκος για κάτι το οποίο δεν είναι νομικά προσδιορισμένο και δεν έχει διεθνώς αποδεκτή σημασία. Ο ορισμός ο οποίος προτείνεται θα έλεγα χρησιμοποιεί αφηρημένους όρους όπως άδικη μεταχείριση ε, και άδικη αντιμετώπιση των εργαζομένων. Κοιτάξτε, η αδικία είναι κάτι το πολύ υποκειμενικό. Αυτό το οποίο είναι άδικο για μένα μπορεί να είναι δίκαιο για κάποιον άλλον. Κάθε επιχείρηση μπορεί να πιστεύει ότι είναι άδικο μια άλλη επιχείρηση να τα καταφέρνει καλύτερα και κάθε εργαζόμενος μπορεί να πιστεύει ότι είναι άδικο ο μισθός του να είναι χαμηλότερος από το μισθό του διπλανού του. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την παραδεχθούμε. Ήμουν λοιπόν λίγο φιλοσοφική σε αυτά που είπα, αλλά σας καλώ να είσαστε πιο πραγματιστές σε αυτά που λέτε εσείς. Ευχαριστώ κύριο Σιλικιώτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον Γιώργο Μπάλα για την όλη καλή δουλειά που έγινε μέχρι σήμερα. Ε, όπως έγινε ξεκάθαρο, οι διεργασίε για συμφωνία και κοινέ τροπολογίε φάνηκε να είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Εμεί είμαστε ικανοποιημένοι για τη δουλειά που έχει μέχρι σήμερα, αλλά λυπόμαστε για τη στάση ορισμένων ομάδων που δυσκολεύουν τη δουλειά του να βγει η έκθεση, για να μην πω ότι ενδεχομένω να υπάρχει και η προσπάθεια για να τραπεί αυτή η εκθεσή και εγώ δεν έμαθα να μασώ τα λόγια μου, θέλω να μιλώ ειλικρινά. Βρεθήκαμε πολλέ φορέ να, συζητούμε ήδη συμφωνημένε τροπολογίε και να απαλαμβάνουμε συχνά τέτοια πράγματα. Κάτι που κάνει τη δουλειά μα ιδιαίτερα μακροχρόνια. Και επειδή ακούω απόψει εδώ ότι βεβαίω ο κόσμο είναι άδικο και πρέπει να τον παραδειχτούμε, καταλαβαίνω ότι κάποιε ομάδε μπορεί να δίνουν μεγάλη σημασία στι δυνάμει τη αγορά και τη δίθεν ανταγωνιστικότητα, αλλά εμεί είμαστε την Επιτροπή Απασχόληση εδώ και Κοινωνικών Υποθέσεων και είμαστε υπόχρεοι πρώτα-πρώτα να στηρίζουμε του εργαζόμενου και βεβαίω με τη στάση μα και τι εκθέσει μα να αλλάζουμε τα δεδομένα και όχι να αποδεχόμαστε πραγματικότητε. Εμεί στηρίζουμε την προσπάθεια που γίνεται σε αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση παραμένοντα προσιλωμένοι στι αρχέ μα. Δηλαδή, ποιε πρέπει να είναι οι αρχέ μα προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τη ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτου, τη καταπολέμηση του κοινωνικού κάμπινγκ, το οποίο επιτελείται για χάρη τη δίθεν ανταγωνιστικότητα, στην, στην πραγματικότητα όμω τι, τι α... επιτελείται υπέρ τη ασίδωτη κατά την άποψή μα κερδοφορία των εταιριών σε βάρο των εργαζομένων. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που εμεί στηρίζουμε όλε εκείνε τι συμβαστικέ οι οποίε υπογραμμίζουν την ανάγκη στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων και όταν μιλούμε για εργασιακά δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται και οι συλλογικέ συμβάσει και το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση. Και όχι ε, τα ατομικά συμβόλαια, τα συμβόλαια που καταργούν εργασιακά δικαιώματα που κερδίθηκαν με ε, αγώνε δεκάδων ε, χρόνων των εργαζομένων. Θεωρούμε μάλιστα ότι η έκθεση πρέπει να αποτελέσει μια δυνατή φωνή του Κοινοβουλίου υπέρ των εργαζομένων ενάντια στις πολιτικές απορρίθμισης των μισών και των δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα αυτή τη χρονική στιγμή όπου συζητείται η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και ναι, αγαπητοί συνάδελφο στο Φιλεθέρο, ναι, είμαστε υπέρ των ίσων δικαιωμάτων τη ίση αμοιβή για την ίση συνεργασία. Και αυτό είναι που πρέπει να παλεύουμε. Αν καταλαβαίνουμε ότι ναι υπάρχουν αδικίες, αγωνιζόμαστε για να τρέψουμε αυτές τι αδικίες και ιδιαίτερα αυτό που προσπαθεί και διαφημίζει σήμερα η, η Κομισιόν για το κοινωνικό τριπλό A. Ε, θέλω να επαναλάβω ότι ε, εμεί ω ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, της Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, σα στηρίξουμε ε, τη δουλειά που γίνεται, γιατί πρέπει να βγει μια έκθεση ακριβώς που βασική της αρχή πρέπει να είναι η περάσπιση των εργαζομένων και του κοινωνικού κράτους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η Καρίμα Ντέλ εκ μέρους των Πρεσέντων είναι εδώ. Άρα πάμε στο EFTD και την Λάουρα Άγγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώμ για τη δουλειά που έχει κάνει. Ήταν κάτι το δύσκολο αυτό που έκανε. Το ήξερε ο Γιώμ, από την αρχή και εμεί σήμερα ξέρουμε τι μας περιμένει όταν να περάσουμε στην αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Αυτό το οποίο είναι σαφές μετά από 20 συναντήσεις των σκιωδών είναι ότι οι θέσεις αφίστανται μεταξύ τους και δεν είναι εύκολο να συμβιβαστούν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι ε, για τη δική μου ομάδα για να υποστηρίξει την πρόταση του Γκυγιόν Μπαλάς είναι κάτι το δεδομένο. Από την άλλη βέβαια κατανοώ τις ανησυχίες των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων. Έχουμε διαφορετικά παρελθόντα θα έλεγα και πλαίσια ο καθένας και ο καθένας θέλει να υπερασπιστεί τα ειδικά χαρακτηριστικά της δικής του χώρας. Ακούσα κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα έλεγα αναφέρθηκαν σε πολύ σημαντικά και θεωρητικά θέματα. Αυτό δεν είναι κριτική αλλά Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και αυτό δεν είναι εύκολο. Είναι όμως προφανές ε, ποιες είναι οι οικονομικές συνθήκες που κρατούν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που με τη σειρά τους καθορίζουν την προβληματική αντιμετώπιση ε, των σημαντικών προβλημάτων που επηρεάζουν τις διάφορες χώρες. Συνεπώς ε, θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση γιατί εμείς στην Ευρώπη αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε κάποιες προκλήσεις ε, και κάποιες επιλογές οι οποίες θα έχουν σημαντικότερες επιβαρύνσεις θα επιφέρουν στο μέλλον. Γιατί σήμερα μιλάμε για το κοινωνικό ντάμπινγκ στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκεφτείτε τι θα πρέπει να κάνουμε αν δούμε το τι γίνεται με τον τρόπο που επηρεάζουν άλλες οικονομίες, άλλες οικονομικές πραγματικότητες στην δική μας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι δεν ξέρω αν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή ε, να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Μήπως θα έπρεπε να προηγηθεί η αναθεώρηση της οδηγίας είναι σαφές ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλήρως ότι αντιπροσωπεύουμε 28 χώρες, 28 διαφορετικές πραγματικότητες, όπου ο ανταγωνισμός δεν είναι θεμητός πάντα, όπου δεν υπάρχουν οι ίδιες εγγυήσεις για τους εργαζομένους και οι κοινωνικές εγγυήσεις και όχι μόνο στα εργασιακά ειδικά, και νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο βγαίνει στην επιφάνεια είναι μια τεράστια δυσκολία να συμβιβαστούμε. Α συνεχίσουμε λοιπόν τις συζητήσεις, ας συνεχίσουμε να το εξετάζουμε το θέμα και να προετοιμάσουμε θα έλεγα κυρίως την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Αυτό θα είναι κάτι το περίπλοκο ε, θα έχουμε δύο εισήγητές οι οποίοι εκινούν από δύο διαφορετικές θέσεις και αυτό ε, θα πρέπει να μας οδηγήσει στο τι είναι δυνατόν να γίνει γιατί μπορούμε να λέμε τα ίδια και το αντίθετό του στην ίδια ακριβώς στιγμή. Ευχαριστώ κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Μπάλας, όμως έχω ένα προβληματάκι ε, για ένα μικρό θέμα ε, σχετικά με το, αυτό που είπε ο κύριος Μπάλας. Ε, η τελευταία επιτροπή σχετικά με την έκθεση των Μπένσκι, είχε κάνει μια προετοιμασία, όμως τότε η συγκεκριά ήταν η κυρία Μποϊζότο και ο κύριος Μπάλλα είχε ξεκάθαρα αρνηθεί όλα τα συμβιβαστικά κείμενα να μεταφερθούν στην κυρία Μποϊζότο. Αυτό που μας εκπλήσει ακόμα περισσότερο, κυρία Πρόεδρε, γιατί θέλω να είμαι λίγο πιο ισχυρό στις απόψεις μου, είναι ότι η γραμματεία της Επιτραπής τελικά υπέξει στον κύριο Μπάλλας. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα συγκεκριμένο συζητητής ε, ε, θα πρέπει ε, να κάνουμε αυτό που λέει ο κύριος Μπάλα, ο οποίος απευθύνθηκε στη γραμματεία για να μην μεταδώσει τα κείμενα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο δημοκρατικοί. Και τώρα λέει ότι είναι χαρούμενος και θα κάνει τα πάντα για να μπορέσει να έχει μια κοινή, να έχουν μια κοινή θέση όλοι οι αιρετοί. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολιτική που δεν αποδεχόμαστε και νομίζω ότι εδώ ε, θα είμαι πιο έξυπνο από τον κύριο Μπάλλας, γιατί ε, συμμερίζομαι αυτό που λέει όταν λέει ότι το κοινωνικό dumping και η έκθεση γι' αυτό δεν θα πρέπει να μιλά για το θέμα των αποσπασμένων. Να πω στον κύριο Μπάλλας και στους υπόλοιπους της Επιτροπής ότι είμαι σίγουρος ε, πως η αναθεώρηση της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους που τόσο πολύ μας απασχολεί, ήσυχα και σταθερά θα θαυτεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you. Ευχαριστούμε. Αυτό σημαίνει ότι πάμε τώρα σε όσους έχουν ζητήσει να μιλήσουν αν μπορείτε, παρακαλώ, για δύο λεπτά ο καθένας. Η κυρία Σατιέ πρώτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ με την ε, σειρά μου, όπως και όλοι οι σκιώδεις, ε, θα ήθελα να χαιρετήσω τον δουλειά που έχει κάνει ο κύριος Μπάλας ως τώρα, να πω όταν έχουμε ε, μια συνάντηση των σκιωδών. Συνήθως ε, κάτι δεν πάει καλά όταν είμαστε λίγοι και γι' αυτό πρέπει να το προσέχουμε ιδιαίτερα. Εδώ είναι θέμα μεθόδου νομίζω το πρόβλημα. Βλέπω ότι είναι μεγάλη ο πειρασμός να μιλάμε για την αναθεώρηση της οδηγίας των αποσπασμένων, ενώ έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτή η σύγχυση στην ουσία μας οδηγεί ε, στο να έχουμε υπέρμετρες προκλήσεις ε, που διακυβεύουν ουσιαστικά το ίδιο το θέμα της εργασίας μας. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Το δεύτερο είναι ότι όταν αφινόμαστε σε αυτό, τι γίνεται, ε, εκ των προτέρων κάνουμε πιο πολύπλοκη την αναθεώρηση της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό το παιχνίδι. Το είπατε ότι υπάρχουν διάφορες πολιτικές απόψεις, ε, μιλάμε συνεχώς για πολιτικές ομάδες, ε, που ε, κάποιες φορές ε, ε, έτσι όπως τίθεται το θέμα, φαίνεται τη μία ότι είναι τα κρατημέλη, την άλλη πολιτικές ομάδες που έχουν το ζήτημα και τελικά είναι δύσκολο να βρεθεί η συνένεση. Όταν ε, περιχαρακωνόμαστε σε τέτοιες θέσεις, λοιπόν, μπορεί να έχουμε και 20 και 40 συναντήσεις των συντονιστών, όμως τελικά ό,τι και να γίνει η κατάσταση παραμένει πολύπλοκη. Και εγώ δεν θέλω να θάψουμε αυτή την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Σας το εγγυώμαι ότι δεν θα τη θάψουμε. Απλώς ε, διαφορετικά θα προσεγγίσουμε το θέμα, γιατί σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, όμως ο καθένας έχει την ευθύνη του και πρέπει να βρούμε πού ακριβώς θα συνενέσουμε. Αυτός είναι και ο λόγος ε, που υπάρχουν κάποιοι συμβιβασμοί οι οποίοι, οι οποίοι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά εκείνοι οι συμβιβασμοί που άπτονται άμεσα των επερχόμενων διαπραγματεύσεων για την αποσπασμένη εργασία και συγκεκριμένα μιλάω για τη συμβαστική M, εγώ ως και η Αγνές Γιούγκερ θα ε, πει το ίδιο φαντάζομαι και αυτή ως συνεισηγήτρια για τους ε, αποσπασμένους, σας λέω ότι σφάλετε. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας, ίσως να μην καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο, αλλά αν υπάρχει πραγματικά θέληση να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα των αποσπασμένων, θα πρέπει η έκθεση πρωτοβουλίας ε, για το κοινωνικό dumping να ασχολείται μόνο με αυτό και όχι με άλλα πράγματα. Εγώ θέλω να πω στον κύριο Μπάλλας με την ευκαιρία. Δεν θέλω αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας ε, να υποσκάψει την αναθεώρηση της οδηγίας που είναι απαραίτητη και ε, δεν είναι σε αυτό το διάμεσο διάστημα ε, θεμητό να κάνουμε τέτοια πράγματα και να υποσκάπτουμε το έργο των συνεισηγητριών πρέπει να, θέλουμε, να ξέρουμε τι θέλουμε με το κοινωνικό dumping. Αν θέλουμε πραγματικά ως Επιτροπή Απασχόλησης να κάνουμε τη δουλειά μας, ας μην αρχίσουμε να τα συγχαίουμε όλα και ας σεβόμαστε κάθε φορά το θέμα της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Κόχ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύνταμος. Ε, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Να πω όμως ότι ε, τα αποτελέσματα της εργασίας των, ε, της Επιτροπής Μεταφορών με τέσσερις συμβιβασμούς είναι πολύ καλά και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Μεταφορών και τον κύριο Μπάλλας για αυτή την πολύ καλή έκβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω η εργασία που έγινε για αυτήν την έκθεση ε, πρωτοβουλίας και οι προτάσει του κυρίου Μπάλας είναι ενδιαφέρουσε, Άκουσα την κυρία Λωράν Σαρτιέ που είπε ότι οι αρχικές προτάσει ήταν άκαμπτες. Ήδη εγώ αρχικά βρίσκω ότι είναι προτάσεις ευρύτατες οι οποίες περιλαμβάνουν Ίσως είναι ο τρόπος ε, κατανόησης. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό, δεν το είπα αυτό, δεν το είπα αυτό. Όχι, όχι, όχι, όχι. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας που να είναι η ευρύτερη δυνατή για τις πρακτικές αθέμη του ανταγωνισμού για τους εργαζόμενους. Αναφέρονται πολλές πρακτικές αθέμη του ανταγωνισμού, οι εταιρείε γραμματοκιβώτιο, το θέμα της αμοιβή, της προστασίας των εργαζομένων αλλά και των αθέμητων παράνομων πρακτικών σχετικά με την αμοιβή των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη έκθεση, αλλά να ζητήσουμε η έκθεση ε, για την καταπολέμηση των αθέμητων πρακτικών να μην περιλαμβάνει το θέμα της οδηγίας περί απόσπασης είναι σαν να ζητούμε να δουλέψει κανείς για την φοροδιαφυγή χωρίς να ασχοληθεί με τους φορολογικούς παραδείσους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την απόσπαση. Νομίζω ότι η οδηγία αυτή θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης μπάλας. Βεβαίως δεν χρειάζεται να μπούμε ε, στις λεπτομέρειες της οδηγίας, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να εντάξουμε το θέμα αυτό. Και σε σχέση με τόσα λέχθηκαν από τη συνάδελφη, παρόλο που η απόσπαση αντιπροσωπεύει μόνο 1% της, του συνόλου των εργαζομένων στην Ευρώπη. Αλλά αν δούμε αναχώρα και ανατομέα τι αντιπροσωπεύει το θέμα της απόσπασης και του αθέμητου ανταγωνισμού που αντιπροσωπεύει, είναι νομίζω σε ορισμένες χώρες μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το 20% με πρακτικές που είναι τελείως αθέμητες, παράνομες και όταν ε, λένε ότι αυτό εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα, αλλά ε, νομίζω ότι οι οικοδομές είναι εσωτερικός τομέας, δεν είναι κάτι που εξάγεται. Θέλετε λοιπόν να έχουμε πρακτικές αθέμητου ανταγωνισμού μέσα στην Ευρώπη που ευνοούν αυτό. Εγώ άκουγα την Ευρώπη και νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες το εννοούν ως μια Ευρώπη που αν είναι αληθές έχει διαφορές στο επίπεδο των κρατών μελών ως προς την κοινωνική προστασία, στόχος μας δεν είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα, αλλά αύριο να πάμε σε μια Ευρώπη που προσφέρει περισσότερη και όχι λιγότερη κοινωνική προστασία και αν σήμερα υπάρχουν διαφορές, θα πρέπει οι διαφορές αυτές να πηγαίνουν προς περισσότερη προστασία και όχι προς λιγότερη. Έτσι εγώ αντιλαμβάνομαι ε, την Ευρώπη όταν μιλάμε για για διαφορές, διχογνωμίες. Θα ήθελα να οδηγηθούμε προς περισσότερη προστασία, όπως ο κύριος Μπάλας, με μηχανισμούς που θα τίνουν προς αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριος Καλισόμπο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά εφόσον ο εισηγητής είναι της γλώσσας του Μολιέρου και θα πω πρώτα απ' όλα ότι υποστηρίζω τα όσα λέχθηκαν από τη συνάδελφο Νταλή, Μαρτίνα και μιλώ εγώ προσωπικά και όχι εξ ονόματος ε, της ομάδας. Αντίθετα με τα όσα είπε η Λάουρα Εχέα, θα ήθελα να τα δούμε αυτά από ευρωπαϊκής απόψεως και όχι εθνικής. Και διαμέσου μιας θεώρησης πολιτικής. Θαυμάζω την εργασία που έγινε. Ξέρω πόσο ήταν δύσκολη, το έζησα διαμέσου της Μαρτίνα και η ομάδα μου συνεχώς έπρεπε να παρακολουθεί την εργασία αυτή, αλλά δεν είναι επειδή έγινε μια σκληρή εργασία το αποτέλεσμα ε, να είναι το πιο ικανοποιητικό μπορούσαμε να κάνουμε κάτι το περίπου ιστορικό, δηλαδή να δώσουμε τον ορισμό του κοινωνικού dumping. Δεν μπορούμε να το κάνουμε δημιουργώντας τέσσερους άλλους ορισμούς τελείως αυθαίρετους, όπως το disempay, όπως είναι η social fraud. Τι είναι η social fraud, υπάρχουν κανόνες, είμαστε κράτη δικαίου νομίζω, όπως είναι η unfair competition, ο αθέμητος ανταγωνισμός, ε, τι είναι, τι είναι αυτό. Και όπως είναι το equal pay, δηλαδή ίση αμοιβή για ίσια εργασία, ε, ίση θέση και ίσο μέρος. Σε ε, μια επιχείρηση βάζετε δύο άτομα που είναι αντιπρόσωποι εμπορικοί, θα κερδίσουν διαφορετικά το ίδιο χρόνο. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά πρέπει πρωτού χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια αρχή να δώσουμε τον ορισμό για να μην χειραγωγείται. Βεβαίως γίνεται μια αναφορά σε κατηγορίες ατόμων, ε, σε ε, ε, κάποιον αναλογιστής που εντάσσεται στις συλλογικές συμβάσεις. Αλλά όλα αυτά πρέπει να προσδιοριστούν το να λέμε αυτά μας οδηγούν σε αντιπαραθέσεις που δεν θα κάνουν την Ευρώπη να προοδεύσει για το καλό του εργαζομένου του Ευρωπαίου. Αισθάνομαι πολύ άσχημα με το κείμενο αυτό και δεν θα υποκύψω. Πρώτα πρέπει να προστατεύσουμε την ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα, όχι για το 1% ή το 20% για όλους, αλλά να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό για του κόστου εργασίας, διότι στην Ισπανία, στην δική μου εκλογική περιφέρεια, μπορέσαμε να βγούμε από την Άβυσσο χάρη στον ανταγωνισμό ε, διαμέσα στο κόστος εργασίας, διαμέσου του κόστου εργασίας. Και νόμιζα ότι αυτό θα εξεταζόταν, να υπάρχουν ελάχιστοι κανόνες ε, κοινωνικοί, απαιτητοί για όλους τους πολίτες, για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό συμφωνώ ενώ για όλους θα έχουμε ίσους όρους, θα έχουμε ελάχιστα κοινωνικούς κανόνες, πρέπει να αφήσουμε τις δυνάμεις της αγοράς να ε, λειτουργήσουν. Όταν μιλούμε για αποσπόμενους εργαζόμενους, πρέπει να πω κάτι. Ή λαμβάνουμε την απόφαση να έχουμε μία μόνη παράγραφο που λέμε ότι τα προβλήματα του κοινωνικού dumping αντικατοπτρίζονται στους εργαζόμενους που διαβαίνουν τα σύνορα και, και ότι θα, το... Θα, το... ασχοληθούμε με το ψήφισμα το επόμενο ή κάνουμε την εργασία μας για το κοινωνικό ντάμπινγκ όταν η κυρία Λόραν Σαρτιέ και οι συνάδελφοί της θα τελειώσουν την εργασία τους. Αλλά δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την εργασία εδώ, δεν μπορούμε να την ορίσουμε εδώ αυτήν την εργασία. Είναι θεωρητικά επικίνδυνο. Ή κάνουμε ε, για, το, ε, για τους εργαζόμενους τους αποσπόμενους και μιλάμε για αυτό που είναι πραγματικά ένα πρόβλημα ή προσπαθούμε να έχουμε μια έκθεση και εγώ μιλάω ως πολιτικός και καταλαβαίνω πολύ καλά τους συναδέλφους μας ή έχουμε μια έκθεση για να ικανοποιήσουμε ένα πρόβλημα πολιτικό πάρα πολύ συγκεκριμένο σε ορισμένες χώρες. Και εδώ τους λέω κάτι. Μην θυσιάστε την κινητικότητα των εργαζομένων σε μια ανάγκη πολιτική και ε, μην προσπαθήσετε ένα αντίγραφο να το κάνετε, ένα πρωτότυπο ε, που δεν ικανοποιεί. Αν θέλουμε την κινητικότητα ε, για, να αποφύγουμε τον λαϊκισμό και τον ρατσισμό, όχι. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα μικρό πράγμα που θα είναι δίθεν, κατά τη γνώμη μου. Και τελικά δεν καταλαβαίνω, εξακολουθούμε να παραπέουμε λίγο, αξιολογούμε τις ε, κανόνες εργασίας ε, που μας έφερε η Επιτροπή Μεταφορών, αλλά ξέρετε πόσα άρθρα θα μπορούσα να σας προτείνω για τον τουρισμό, για τη γεωργία, για την άμυνα, όπου προσλαμβάνονται με υπεργολαβίες, με προστασίες λιγότερες για τους νέους που θα πάνε να πεθάνουν εκεί στο Αφγανιστάν. Και αυτό είναι κοινωνικό ντάμπινγκ επίσης γιατί κάνουμε ένα μέγα κείμενο όπου καλύπτουμε όλα και τελικά δεν καλύπτουμε το κοινωνικό dumping, το ουσιώδες. Έχω πάρα πολλές δυσκολίες με αυτό το κείμενο όπως έχει τεθεί τώρα. Θα ήθελα να επανέλθουμε, όπως είπε η κυρία Σαρτιέ, στην ουσία το προβλήματος ε, και να ε, περιχαράξουμε τις αντιλήψεις χωρίς να έχουμε ιδεολικούς όρους ασαφείς. Ε, για ψηφοθυρικούς λόγους. Θα κερδίζαμε πολλά. Εγώ προσωπικά δεν μιλάω εξ ονόματος της ομάδας, η Μαρτίνα μιλάει εξ ονόματος της ομάδας. Εγώ δεν βρίσκω τη σαφήνεια και την ποιότητα επαρκή για να μπορέσω να ψηφίσω το κείμενο αυτό. Thank you and uh, try to stick. Ευχαριστώ. Προσπαθήστε παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο σας γιατί θα πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Μαν. Δεν είναι απλό ε, να μας το ζητάτε αυτό, γιατί ο προηγούμενος έπρεπε να μιλήσει δύο λεπτά και μίλησε εξήμιση. Ξεκινάμε λοιπόν ε, ε λέγοντας ότι είχαμε 18 λεπτά καθυστέρηση ξεκινώντας αυτή τη συνεδρίαση, οπότε ε, θα πρέπει κάπως να προσπαθήσουμε να συμβιβαστούμε και σε αυτό. Αυτό που είπε ο Γκυγιώμη ήταν πολύ σημαντικό. Έγιναν πολλές συζητήσεις με τους σκιώδεις ε, και το να έχουμε 20 τέτοιες ε, συνεδριάσεις είναι ένα μικρό ρεκόρ για μια τέτοια έκθεση. Νομίζω θα πρέπει τουλάχιστον να θίξουμε το θέμα των αποσπασμένων, όμως ε, να μην κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα μπορέσουμε μετά να τηρήσουμε ε, πρέπει να δούμε οπωσδήποτε τι γίνεται με τις πρακτικές των αποσπασμένων. Να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν κοινό ορισμό, ο οποίος ε, θεωρώ ότι θα ήταν κάτι σωστό για να μην ε, υπάρξουν μέτρα καταχρηστικά. Δεύτερον, επίσης υπάρχει η οικονομική πτυχή. Θεωρώ ότι είναι σωστό να δούμε τι γίνεται όταν μιλάμε για στρέβλωση της αγοράς και για τις ανισότητες. Υπάρχουν οι κοινωνικές πτυχές, είναι αυτό που εμείς κάνουμε ακριβώς. Προσπαθούμε να δούμε τις επιπτώσεις, να δούμε ε, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια, ένας ορισμός καλό θα ήταν να υπάρχει. Ο ορισμός που έχει ήδη βρεθεί είναι πάρα πολύ περίπλοκος και δυσκολεύει την έβρεση υποστήριξη. Νομίζω επίσης ότι για το θέμα των εταιριών βιτρίνα ε, είναι πολύ σημαντικό να το θίξουμε, να δούμε και την ε, ε, προσωρινή εργασία, αλλά να μην έχουμε μία έκθεση μόνο για αυτή. Θα πρέπει να την ενσωματώσουμε και στις υπόλοιπες τέτοιε που κάνουμε για την ευκαιριακή απασχόληση, εκθέσει που κάνουμε για την ευκαιριακή απασχόληση και έτσι, έτσι ώστε να δούμε ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των ε, εργαζομένων που πλήττονται από αυτό. Επίσης, θα ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα που μπορεί να προκύψει στο ΕΛΚ είναι το θέμα της αναλογικότητας, ναι, αυτονόητο, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Θα ήθελα να έχουμε ένα ελάχιστο έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η συζήτηση, γιατί νομίζω ότι απέχουμε από αυτό. Και τώρα αν χρειαζόμαστε 20 πάλι συνεδριάσεις, δεν ξέρω. Ε, αν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Ιούλιο, 13 Ιουλίου θα τα έχουμε καταφέρουμε Ίσως ε, θα πρέπει να αναβάλουμε κάτι άλλο έτσι ώστε ε, την επόμενη φορά που θα γίνει η προσπάθεια τη Δευτέρα του Στρασβούργου να ασχοληθούμε ε, σύντομα με κάποιες εκθέσεις να μην γίνει γιατί χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη και εντελεχή συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Ε, νομίζω ότι με τα τρία λεπτά είμαι λίγο πολύ κοντά σε αυτό που ζήτησε η Πρόεδρος. Να μιλήσουμε δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Mann, for... Ευχαριστώ κύριε Μαν για τα τρία λεπτά. Ήταν ακριβώς αυτό που είπατε ότι όλοι ε, θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν σύμφωνα με την σειρά που έχουν στον κατάλογο, αλλά θα πρέπει να είναι σύντομοι γιατί θα αργήσουμε για την επόμενη συνεδρίαση. Παρ' όλα αυτά αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για μας και πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Η κυρία Σοφία Ρουμπέιρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις ε, για τη μεγάλη αφοσίωση που έδειξαν για αυτό το θέμα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να παρεκτραπούμε από την ουσία του ζητήματος. Όταν επικεντρωνόμαστε μιλώντας ε, για το social dumping στους αποσπασμένους εργαζόμενους, στην ουσία ξεχνάμε άλλα είδη και δεν ξέρω αν αυτό γίνεται θελημένα ή όχι, ε, άλλα είδη ε, παρέκκλησης από, τα, ε, από τις ελάχιστες συνθήκες που θα έχουν, πρέπει να έχουμε διασφαλίσει. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, σε ανθρώπους αυτοαπασχολούμενους ε, υποτίθεται που χρησιμοποιούνται τελικά ως ε, υπάλληλοι. Υπάρχουν δάσκαλοι στην Πορτογαλία που παίρνουν ε, ε, την ε, άδεια να δράσουν ως αυτοαπασχολούμενοι στην Πορτογαλία όπως γίνεται, αλλά δεν είναι αυτοαπασχολούμενοι. Θα πρέπει λοιπόν να συντονιστούν οι επιθεωρήσεις εργασίας στα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σωστό επίπεδο προστασίας. Δεύτερον, όταν μιλάμε για το κοινωνικό dumping θα πρέπει να προσέχουμε, διότι είναι αυτό μία περίπτωση ε, όπου, ε, ε, σύμφωνα με την οποία η ανταγωνιστικότητα βασίζεται ξεκάθαρα στο κόστος στο μισθολογικό, ενώ η ανταγωνιστικότητα θα έπρεπε να προέρχεται από την προστιθέμενη αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της στους πολίτες. Άρα, το θέμα συζήτησης είναι ευρύτερο και έχει να κάνει με την ανάπτυξη που επιθυμούμε για την Ευρώπη. Να σας θυμίσω τέλος ότι η ίδια η Επιτροπή Υπεραμήνθηκε της ε, ισχύω του κοινωνικού πυλώνα και αναφέραμε στον κύριο Μαν που είπε ότι χρειαζόμαστε ένα ελάχιστο πλαίσιο για να πατάξουμε το κοινωνικό ε, dumping και ότι χρειαζόμαστε σύγκληση ε, ως προς τα καλύτερα κοινωνικά στάνταρ. Να μην ξεχνάμε όμως ότι αυτή η σύγκληση έχει άλλες επιπτώσεις ε, που έχουν να κάνουν με τη μεγαλύτερη οικονομική και χρηματοπιστωτική σύγκληση. Χωρίς τη δεύτερη δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνική σύγκληση, γιατί αλληλοσυνδέονται τα δύο αυτά στοιχεία. Και πραγματικά, συνάδελφοι, το να μην ε, ε ασχολούμαστε με τις εταιρείες και με τα κράτη-μέλη ε, δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σαν να είναι άμυρα ευθυνών και αυτά, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε την σύγκληση. Ευχαριστώ. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, Πρόεδρε, από αυτά τα οποία ακούγονται. Αυτοί που δεν ξέρουν τι σημαίνει ίση απασχόληση, ίση αμοιβή, να τους παραπέμψω στη σταθερή ευρωπαϊκή νομολογία που έχει καταδικάσει πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες μέλη, γιατί πράγματι διαφοροποιούσαν την κατάσταση μισθολογικά, ενώ οι εργαζόμενοι έκαναν την ίδια δουλειά. Τώρα αν είναι βλάκες οι ευρωδικαστές αυτό είναι άλλο θέμα, τίθεται ίσως κάποιοι άλλοι να είναι βλάκες και εδώ στην αίθουσα. Πάντως είναι σαφές ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί έχω την εντύπωση ότι για πολύ καιρό οι ευρωβουλευτές δεν είχαν την ίδια αμοιβή και τα εναρμονίσαμε όλα είτε είστε από τη Μάλτα, είτε είστε από τη Σουηδία, τώρα έχουμε όλη την ίδια αμοιβή. Ενώ δεν συνέβαινε αυτό. Οπότε κάποιοι έχουν και πιστεύουν στην αρχή ίση απασχόληση, ίση εργασία, εναρμόνιση λοιπόν. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε διαφορετικοί, μπορούμε να σεβόμεθα την πολλαπλότητα, αλλά να σεβόμαστε ο ένας την εργασία του άλλου. Υποστηρίζω λοιπόν την προσπάθεια που κάνει ο Κιγιόν Μπαλάς γιατί οι εργαζόμενοι συμμερίζονται τις απόψεις του Μπαλάς. Και αν πράγματι σε επίπεδο αριθμών αυτό δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν εκατομμύρια αποσπόμενοι εργαζομένοι και οι συνέπειες στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων είναι τεράστιες. Ας φανταστούμε ότι αύριο και αυτό φοβάμαι θα συμβεί γιατί νομίζω ότι η συζήτηση που θα γίνει είναι ότι η ανταγωνιστικότητα των κρατών δεν πρέπει να γίνεται μόνο μέσα από το κόστος της εργασίας. Ας φανταστούμε αύριο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει την οικονομία, το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς ε, για την Κίνα. Τότε οι Κινέζοι θα συμφωνήσουν όλοι ότι μόνο το κόστος της εργασίας μετράει. Ευχαριστώ η κυρία Γιασοβιέσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζήτησα για μια ακόμη φορά το λόγο γιατί μερικές φορές οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται στην Επιτροπή μας με εκπλήσουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες των νομοθετικών μας ενεργειών, όχι μόνο για σήμερα και αύριο, αλλά μακροπρόθεσμα να προσπαθήσουμε να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει η νομοθετική μας δραστηριότητα στους διάφορους τομείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα επηρεαστούν από τα μέτρα τα οποία εμείς ψηφίζουμε. Από ό,τι μου φαίνεται λοιπόν, είμαστε λίγο χαλαροί και λίγο πρόχειροι με τον τρόπο με τον οποίο ε, θέλουμε να εκδίδουμε συστάσεις και πολλές φορές οι συστάσεις αυτές είναι μονόπλευρες. Και δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις, τις αρνητικές φυσικά, των συστάσεων αυτών. Θα πρέπει να δούμε και τις άλλες επιλογές, θα πρέπει να δούμε τα συν και τα πλήν. Θα πρέπει να δούμε το ποιοι θα ε, αποδεχθούν κάποιες επιλογές και ποιοι όχι. βέβαια αυτή τη διαδικασία την αναλυτική δεν την κάνουμε πάντα όταν συντάσσουμε συστάσεις στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δυστυχώς η προσπάθεια την οποία εμείς κάνουμε θα πρέπει να έχει σαν στόχο η νομοθεσία που προτείνουμε να είναι ξεκάθαρη και διαφανής. Και δυστυχώς στις εκθέσεις που υιοθετούμε δεν ισχύει πάντα κάτι τέτοιο. Να πω κάτι για την κυρία Αρενά ε, στην αρχή της συζήτησης πολλές πολιτικές ομάδες είχαν προτείνει την ομάδα ε, ε, κάποιων συμβιβαστικών τροπολογιών γενικότερα για το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων, γιατί το κοινωνικό ντάμπινγκ τους αφορά φυσικά. Αλλά δεν θα πρέπει να παρερμηνευθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ σαν κάτι που έχει σχέση μόνο με τους υποαπόσπαση εργαζομένους. Γι' αυτό ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε να προτείνουμε σε πάρα πολλά σημεία της έκθεσης, να μην πω πάνω από δέκα παραγράφους, αναφερόμαστε συστηματικά στην απόσπαση των εργαζομένων. Η πολιτική μας ομάδα έχει αποφασίσει ότι αυτή δεν είναι δική μας δουλειά υπάρχει μια έκθεση για την απόσπαση των εργαζομένων, θα πρέπει να σεβαστούμε την προσπάθεια που κάνουν οι συνάδελφοι και δεν θα πρέπει να ανακατευτούμε εμείς με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαλάς, να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις για την προσπάθεια που έχουν κάνει, όπως επίσης και για την προσπάθεια που μένει ακόμη να γίνει για τις συμβιβαστικές προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί. Θα ήθελα να σημειώσω και να χαιρετήσω τον ορισμό του κοινωνικού ντάμπινγκ. Είναι ένας ορισμός ο οποίος σαφώς και θα πρέπει να βελτιωθεί, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα και είναι σημαντικό να καθορίσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο περαιτέρω να επιμείνουμε στο θέμα της μεθόδου, όπως το έκαναν και κάποιοι από τους συναδέλφους. Το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων, των αποσπασμένων ή απόσπαση εργαζομένων είναι σημαντικό για πάρα πολλές χώρες. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, έχει σημασία για τους εργαζομένους και για τις επιχειρήσεις. Έχει σημασία και κοινωνικά και οικονομικά αλλά και πολιτικά σε κάποιες από τις χώρες μας πέραν αυτού για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο χρόνο. Είμαι και εγώ υπέρ του να διακρίνουμε τις συζητήσεις τις οποίες κάνουμε για το κοινωνικό ντάμπινγκ που είναι ένα πραγματικό πρόβλημα ε, στο οποίο πρέπει να κάνουμε βήματα και από την άλλη να αφήσουμε τους δύο συνεισηγητές ε, να προχωρήσουν για τη δική τους υπόθεση, το θέμα δηλαδή της απόσπασης των εργαζομένων. Γιατί ο κίνδυνος είναι να μην καταλήξουμε πουθενά. Ας εργαστούμε λοιπόν για το κοινωνικό ντάμπινγκ, ας δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, το χρειαζόμαστε. Οι διαφοροποιήσεις δεν είναι μόνο εθνικού τύπου, είναι διαφοροποιήσεις και στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων, ιδιαίτερα για τους υποαπόσπαση εργαζομένους. Ευχαριστώ. Ναι, κυρία Πρόεδρε, κύριος Δαντβίλε. Ναι, συμμερίζουμε τα, τις περισσότερες παρεμβάσεις των ομάδων, ε, των εκπροσώπων ε, των, της ομάδας του ΕΛΚ, αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε ένα από τα επιχειρήματα που αναφέρθηκε από τον Εντουάρ Μαρτά, σχετικά με το ίση αμοιβή για ίση εργασία. Πάρουμε το παράδειγμα των ευρωβουλευτών. Εφόσον ε, έχουμε ίση ε, θητεία, ίση αμοιβή, αν ήταν ίση εργασία, ε, για ίση εργασία, ίση αμοιβή, αν λάβουμε υπόψη το, το πώς είναι εδώ παρόντες, δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό, παρόλο που στη Γαλλία λέμε ότι πάρα πολύ συχνά στην ε, λειτουργία ο ιερέας ε, μαλώνει αυτούς ε, που είναι εκεί. Πολύ καλά. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Μπαλάσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ στους συναδέλφους για όλες τις παρατηρήσεις τους. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ στα όσα λέχθηκαν παρόλο που δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σχετικά με τα όσα είπε ε, στην αρχή από τα Σαλέχτιαν ξέρουμε τα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε. Δεν μιλάω για την απόσπαση, εκτός από την απόσπαση των εργαζομένων, όπου υπάρχουν εφικτές πρόοδοι. Το θέμα της αεροπορίας εκεί η Επιτροπή Μεταφορών μας είχε αναφέρει ότι ορισμένα στοιχεία τα οποία εντάξαμε σχετικά με το θέμα, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά το αίτημα. Αλλά για τα υπόλοιπα βεβαίως προσπαθούμε να βρούμε τρόπους που να μπορούν να συμβιβάσουν αυτό το οποίο εσείς υποστηρίζετε και εμείς υποστηρίζουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα σας απαντήσω ταυτόχρονα στην κυρία Τζαμπάλοβα για το θέμα της απόσπασης διότι είναι θέματα της πολιτικής συζήτησης και η κυρία Τζαμπάλοβα έχουμε μια βασική διχογνωμία ε, όπως και με το συναδελφό της, αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Σήμερα οι παράγραφοι των συμβιβασμών που αναφέρονται ουσιαστικά στην αποσπασμένη εργασία είναι 3 ε, από 37. Να πούμε λοιπόν ότι η καρδιά της έκθεσης, όπως το άκουσα να λέγεται, και αναφέρεται στην αποσπασμένη εργασία, είπα κυρίως, κυρίως και ότι μιλάμε ε, για την αποσπασμένη εργασία, δεν είναι μόνο, δεν είναι αληθές και αν πάρετε όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες όπου αναφέρεται το θέμα αυτό, είναι 8 στις 37. Προσοχή λοιπόν να μιλάμε σήμερα ότι η έκθεση αυτή επικεντρώνεται στο θέμα των αποσπόμενων ε, εργαζομένων. Δεν είναι αληθές αυτό. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο σχετικά με τον τρόπο που μπορούμε να εργαστούμε. Εγώ καταλαβαίνω και αυτό λέχθηκε από τον κύριο Καλτεσόμπο... Ε, θα μπορούσαμε να μην εργανιστούμε για την αποσπασμένη εργασία παρά μόνο ε, για την κοινωνική σύγκληση. Πώς θα μπορούσαν τα δικαιώματα να συγκλίνουν. Αυτό κάναμε στο τρίτο μέρος της έκθεσης που είναι αποτέλεσμα της ε, διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις ομάδες όπου μπορούμε να έχουμε το μέγιστο που μπορούμε σχετικά με το θέμα αυτό. Σας διαβεβαιώνω κύριε Σομπό ότι αν μπορούσα να πάω πιο μακριά θα το είχα κάνει αλλά ακόμα και η ομάδα του σχετικά με το σημείο αυτό υπήρξε αρκετά στεναρή, διότι ότι δεν θέλουν να ανοίξουν ορισμένα θέματα. Θα πρέπει να μιλήσουμε ή όχι για το θέμα της αποσπασμένης εργασίας σε αυτή την έκθεση. Προσοχή. Δεν θα μιλήσουμε ποτέ για την αποσπασμένη εργασία αν δεν την αναφέρουμε εδώ. Ας ε, μην το κρύβουμε αυτό, το, την ιδέα να μην μιλήσουμε καθόλου για την αποσπασμένη εργασία σε αυτήν την έκθεση. Δεν είναι για να αφήσουμε την ελευθερία στους συνεισηγητές να μιλήσουν αργότερα για το θέμα αυτό. Είναι επειδή ορισμένοι από εμά και έχουν το δικαίωμα θεωρούν ότι δεν πρέπει να θίξουμε το θέμα αυτό και να μην ξανανοίξουμε την οδηγία του 96 και για το θέμα αυτό ε, ε, άλλαξα πολύ διότι το θέμα της οδηγίας του 96 υπήρχε περίπου σε όλη την έκθεση. Ακολούθησα τις ε, καλές συμβουλές της κυρία Γιασλόβικα για το θέμα αυτό μειώνοντας τις σε δύο βασικές παραγράφους το L και το M διότι εάν η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα στην έκθεση αυτή, τίποτα που να αναφέρεται στην αποσπασμένη εργασία ούτε ως αρχή. Θα ξαναβρεθούμε σε μια κατάσταση όπου για να ανοίξουμε την συζήτηση μετά τη διαδικασία των κίτρινων καρτελών της Κομισιόν δεν θα είναι και τόσο απλό και το επαναλαμβάνω, αυτό που έχετε μπροστά σας, δηλαδή τον συμβιβασμό ΙΒ και τον συμβιβασμό ΙΓ, είναι υποσυζήτηση. Μου είπαν ορισμένες ομάδες ότι ε, ο στόχος δεν ήταν να τα συζητήσουμε, αλλά να τα αφαιρέσουμε από την έκθεση. Άκουσα την κυρία Μωράν Σαρτιέ, η οποία δεν το ζητούσε ακριβώς αυτό, αλλά ζητούσε ότι σε ορισμένα σημεία να επανέλθουμε στο θέμα, αν κατάλαβα καλά, ε, των επιχειρήσεων ευκαιριακής εργασίας, ε, περιστασιακής εργασίας. Πώς μπορούμε ε, να αντιμετωπίσουμε την αποσπασμένη εργασία μεταξύ μας. Περιμένω για αυτές τις δύο παραγράφους, L και M, ΙΒ και ΙΓ, προτάσεις από τις ομάδες για να μου πούν τι θα ήθελαν να τροποποιήσουν στις παραγράφους αυτές, εφόσον δεν έχω λάβει γνώση ε, των προτάσεών τους και κλείνω λέγοντας ότι για το θέμα του ορισμού, ναι, είναι αλήθεια, μπορεί κανείς βεβαίως ο ορισμός αυτός δεν με ικανοποιεί και εμένα, θα πήγαινα πολύ πιο μακριά. Νομίζω ότι για ορισμένους ε, πηγαίνει πολύ μακριά είναι και ευχαριστώ τους και συγητές που εργάστηκαν καλά για να δεχθούν συμβιβασμός δεν μπορεί ένα συμβιβασμό να ικανοποιήσει όλου. και υπάρχει μια αντίφαση στις παρατηρήσεις που έγιναν για το θέμα αυτό, διότι ορισμένοι λένε είναι πολύ γενικό ο ορισμός και πολύ συχνά από την ίδια ομάδα και άλλοι λένε θα έπρεπε να μπούμε περισσότερο λεπτομέρειες για να έχουμε έναν καλύτερο ορισμό. Αν μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για έναν καλύτερο ορισμό, θα βρεθούμε μπρος σε μια μεγάλη δυσκολία για να μπορέσουν να συμφωνήσουν πάνω από 700 ευρωβουλευτές για τον ακριβή ορισμό του κοινωνικού dumping Και καλύτερα, καλύτερα λοιπόν να μείνουμε εδώ σήμερα. Ξέρω ότι η προσπάθεια αυτή δεν ικανοποιεί όλο τον κόσμο και θα κλείσω για δύο σημεία για τους ψευδοανεξάρτητους, υπάρχουν ε, θέματα ε, για τη σχέση με την επιχείρηση, ε, τι είναι ακριβώς ένας μισθωτός, πώς ελέγχεται και είναι ένα θέμα βασικό για τον χρόνο εργασίας. Είναι μια γκρίζα ζώνη ε, της συγκαλυμμένης εργασίας. Έχουμε αποδώσει λιγότερη σημασία στο θέμα αυτό, διότι ήταν όλη η εργασία που είχε γίνει από τον κύριο Πυρίνσκι για τον τρόπο κατά πολέμησης της συγκαλυμμένης εργασίας και μου φάνηκε ότι θα ήταν μια επανάληψη να αναφερθεί αυτό πολλές φορές στην εισήγηση. Κλείνω και συμπεραίνω λέγοντας ότι κατά τη γνώμη μου έχουμε ήδη μια ευρεία συμφωνία για ορισμένα μέρη της εισήγησης αυτής. Υπάρχουν στοιχεία που είναι σημαντικά που θα πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο και το βασικό είναι το θέμα της αποσπασμένης εργασίας. Άλλη μια φορά προτού διαπιστώσουμε μια ασυμφωνία για το θέμα αυτό ως προς τη μέθοδο, εγώ ζητώ να επανέλθουμε στις δύο βασικές παραγράφους σχετικά με την αποσπασμένη εργασία για να δούμε τι είναι εφικτό ή τι δεν είναι όσο προς την γενική αρχή για το θέμα αυτό σήμερα για να μπορέσουμε να την περιλάβουμε ε, στην έκθεση. Δεν πρέπει να, να μην αναφέρουμε το θέμα αυτό ε, θέλω να σας δώσω τη γνώμη μου, αλλά δώστε μου τα κείμενα, δεν μου απαντήσετε, θα τα έχετε εγκαίρως. Συζήτηση μετά. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά όλους και τον κύριο Μπάλασα περισσότερο από όλους. Πρόκειται, είναι το θέμα στην ημερήσα διάταξη, το οποίο συζητούμε για χρόνια και τώρα βρισκόμαστε ε, στα, στη μισά της εργασίας σχετικά ε, για την, το κοινωνικό dumping, την απόσπαση εργαζομένων και αυτό θα μας απασχολήσει στην εργασία αυτή. Νομίζω αρχίσαμε με καλό τρόπο, έχουμε διαφορές, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές απόψεις μέσα ε, Έχουμε θέματα όπου μπορούμε να βρούμε ε, καλούς συμβιβασμούς. Νομίζω ότι ήδη είχαμε μια πολύ ζωντανή συζήτηση και αυτό έδειξε ότι είναι ε, δυνατό να βρούμε έναν τρόπο να προοδεύσουμε και αυτό είναι σημαντικό για αυτό το Κοινοβούλιο, διότι οι ψηφοφόροι θέλουν αποτελέσματα και θα το πράξουμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε με την εικόνα για την οικονομική ανισότητα, την ακρόαση. Αυτό είναι θέμα, μέρος του προγράμματός μας. PHS 3C50 και μετά στις 3 η ώρα θα ξανασυναντηθούμε και πάλι εδώ. Είναι ενοχλητικό όταν ε, ο Επίτροπη αυτή τη φορά, ο κύριος Κατάινεν, έρχεται ε, στην συνεδρίασή μας και είναι, είμαστε λίγοι στην αίθουσα